Bene, Καλή σας μέρα. Να ξεκινήσουμε την πρωινή μας συνεδρία. Πρώτο σημείο στην ημέρησα διάταξη είναι η έκθεση της συναδέλφου Ουρσκοκ. 45 λεπτά έχουμε στη διάθεσή μας ε, για τη συζήτηση του θέματος αυτού. Θα δώσω αμέσως το λόγο στην συντάκτρια κυρία Ουλσκοκ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω σου ειδικά. Η Ήτρα είναι αρμόδια μεταξύ άλλων για ε, να προσθέσουμε μια σειρά από στο ψήφισμα για τα FEE δίκτυα και βεβαίως και η ΔΕΒΕ θα συμβάλλει. Τα ΕΦΗ δίκτυα είναι το σημείο τομής μεταξύ των τεχνολογιών ενέργειας και των ε, ε, τεχνολογιών πληροφορικής. Πρέπει να ενθαρρύνουμε αυτά τα δίκτυα. Αν ε, θέλουμε, για παράδειγμα, να χρησιμοποιήσουμε αποτελεσματικά τις ραδιοσυχνότητες σε όλη την Ευρώπη και την εφή ενέργεια στα πλαίσια του προσεχούς διαδικτύου αντικειμένων, στα πλαίσια λοιπόν αυτά η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλείται να κάνει τα αναγκαία ε, βήματα για να υπάρξει επιτυχημένη και συνεπής ανάπτυξη ε, για τα δίκτυα αυτά. Και θέλουμε να τεθεί ιδιαίτερη έμφαση στα πλεονεκτήματα και τα ωφέλη που τα εφή δίκτυα μπορούν να προκαλέσουν ε, μειώνοντας τις εκκλήσεις διοξιδίου του άνθρακα Επίσης θα μπορέσουμε να μειώσουμε τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και να βελτιώσουμε και τη μεταφορά ηλεκτρισμού. Οι καταναλωτές επίσης μπορούν να προσαρμόσουν την κατανάλωσή τους με τα υφή συστήματα. Μπορούν να χρησιμοποιούν την ενέργεια κατά τη διάρκεια των χρονικών περίοδων της ημέρας όπου είναι φθηνότερη η ενέργεια. Και επίσης μπορούν να ενημερώνονται πληρέστερα για τα ωράρια. Στη συνέχεια τονίζω την επίγουσα ανάγκη να εξυγχρονιστούν τα δίκτυα μεταφοράς ενέργειας, κυρίως μέσα από τα εφή δίκτυα, ούτως ώστε να έχουμε μια καλύτερη δυνατότητα αποθήκευσης και εξισορρόπησης της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, διευκολύνοντας έτσι την παραγωγή και κατανάλωση από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Επίσης, τα μεμονωμένα συστήματα για παραγωγή και αποθήκευση μικρής κλίμακας ε, στη συνέχεια θα μπορούσαμε να επιδιώξουμε διεύρυνση άλλους τομείς όπως ηλεκτρικά αυτοκίνητα ή άλλου είδους προγράμματα για ε, διαφορετικά είδη ζήτησης. Τέταρτον, υπενθυμίζω σε αυτή την έκθεση ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να υπενθυμίσουμε ότι στην συντριπτική πλειοψηφία των σεναρίων ε, για το 2050 δεν θα είναι δυνατόν να ενσωματώσουμε αποκεντρωμένη διανομή εάν δεν αναπτυχθούν τα τοπικά και περιφερειακά ευφυή δίκτυα διανομής. Οπότε είναι σημαντικό για τις ε, τεχνικές εξελίξεις, ε, να προβλέψουμε τις εξελίξεις και γι' αυτό μέσα στο κείμενο τονίζω ότι είναι σημαντικό να γίνουν και απαιτούμε σε επενδύσεις, ε, σε προγράμματα κοινού συμφέροντος στο Ταμείο για την Διασυνδεδεμένη Ευρώπη. Πέμπτον, Τονίζουμε και εδώ ότι τα ΕΦΗ e μεταξύ άλλων προσφέρουν Μοναδική ευκαιρία για την τόνωση της καινοτομίας και μακροπρόθεσμα να αυξήσουν επίσης τις θέσεις εργασίας και κάτι που μπορεί να είναι πάρα πολύ σημαντικό τόσο για την ε, ανάπτυξη μικρομεσαίων επιχειρήσεων αλλά και για τις μεγάλες επιχειρήσεις προωθείται όπως έλεγα η καινοτομία. Σε αυτή την έκθεση προτείνουμε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να κρίνει αν είναι απαραίτητο βάση του τρίτου πακέτου για την οστερική αγορά ενέργειας να κρίνει αν είναι απαραίτητο λοιπόν να ε, καταθέσει πρόταση για την ε, ε, δημιουργία και την ανάπτυξη εφιών δικτύων ηλεκτρικής ενέργειας διότι μπορούν να εμπλακούν πολλοί παίκτες της αγοράς τονίζοντας έτσι και ενισχύοντας τη δυνατότητα συνεργειών και βιώσιμης ανάπτυξης για τηλεπικοινωνίες όπως και για την διανομή ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν χρειάζεται δηλαδή να στοχεύουμε ένα δίκτυο ε, κάθε φορά, μπορούμε να επιδιώξουμε ε, ένα κοινό σχέδιο για διάφορα είδη δικτύων. Τέλος. Τα ευφυή δίκτυα, αναφέρω στην έκθεση μου, δεν πρέπει να επισύρουν επιπρόσθετα τέλη για τους ε, καταναλωτές, αλλά θα πρέπει να είναι προ όφελο τους, ούτω ώστε να καθοδηγούν οι ίδιοι την κατανάλωση ενέργειας και ε, ενδεχομένως και τη δική τους παραγωγή ενέργειας μέσα από τα δίκτυα μικρής κλίμακας. Τονίζουμε επίσης ότι ε, είναι απαραίτητο να είναι αμφίδρομη η επικοινωνία ανάμεσα στους ε, παραγωγικούς φορείς ε, και τους καταναλωτές όπως και σε πολλούς άλλους τομείς είναι σημαντικό να έχουμε ισχυρή προστασία των καταναλωτών. Εξίσου σημαντικό είναι τα κράτη-μέλη αλλά και οι τοπικές και περιφερειακές αρχές να ε, φτιάξουν και να εφαρμόσουν φορολογικά κίνητρα για τέτοιου είδους διανομή ενέργειας μέσα από τα εφή δίκτυα όμως αυτό θα έπρεπε να επαφεί στην αρμοδιότητα των κρατών μελών και όχι τη Ευρωπαϊκή Ένωση, Η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως μπορεί να λειτουργήσει ως κινητήριος δύναμη για την ε, κατασκευή τέτοιων συστημάτων που έχουν ιδιαίτερη σημασία σε περιφερειακό ε, επίπεδο αλλά και έχουν ιδιαίτερη σημασία από πολιτική άποψη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ συνάδελφε Βανίστερόι. Αγαπητοί συνάδελφοι. Από πλευρά του ΕΛΚ ε, να κάνω μερικά σχόλια για αυτήν την θαυμάσια έκθεση. Νομίζω ότι αν εξετάσουμε όλες τις πλευρές που αντιμετωπίζει η πρόταση αυτή, τονίζει τη σημασία των νέων τεχνολογιών, τη βέλτιστη χρήση του ίντερνετ, και ξέρουμε ότι τώρα ξεκινάνε πολλές διαδικασίες σε αυτό το τομέα, άρα αυτή η γνωμοδότηση που στέλνουμε στη Ρέτζη ε, είναι όντως ε, πολύ χρήσιμη και θα πρέπει να εξετάσουμε κάποια σημεία και στα πλαίσια του, των πολιετών δημοσιονομικών προπτικών βεβαίως. Και επίσης ε, το Ευρωπαϊκό Ινστιτούτο για την Τεχνολογία και την Καινοτομία ασχολείται ιδιαίτερα τώρα στα πρώτα χρόνια με, την, ε, με τα θέματα αυτά της ενέργειας και θα ήθελα να ασχοληθεί και με τα ΕΦΗ e δίκτυα το Ινστιτούτο αυτό. Είναι μια πολύ καλή βάση αυτή. Άρα δεν θέτουμε μόνο ε, ερωτήματα και περιμένουμε να λάβουμε απαντήσεις η Ένωση από μια ε, πολύ πρώιμη φάση προσπαθεί να αξιοποιήσει αυτές τις δέσμες ε, γνώσης και καινοτομίας. Θα ήθελα αυτό να ε, περιληφθεί στην έκθεση. Πολύ, στο πολύ εγγύς μέλλον επίσης θα πάρουμε απόφαση για την περαιτέρω εξέλιξη ορισμένων νέων πτυχών της πολιτικής μας για την ενέργεια πέρα από, αυτούς τους, ε, πέρα από αυτές τις δέσμες ε, ανανέωσης και ενέργειας έχουμε και την γνώση υψηλού επίπεδου η γνώση αυτή υψηλού επίπεδου θα μπορούσε να αξιοποιηθεί από τις διάφορες περιφέρειες. Αυτό το συζητήσαμε όταν κάναμε τους τριμερείς διαλόγους για το πακέτο ορίζων. Ε, Τι σημαίνει αυτό. Σημαίνει ότι υπάρχουν φορείς ε, ε, γνώσης που θα βοηθήσουν να εισαχθούν τα ευφυή δίκτυα. Πρέπει όμως να μπορέσουν να εμπλακούν ακριβώς θα πρέπει να αξιοποιήσουμε τα διαφθορτικά ταμεία για να βοηθήσουμε αυτούς τους φορείς. Η γνωμοδότηση λοιπόν αυτή δεν ε, θα είναι χρήσιμη μόνο για τη δική μας την Επιτροπή. Όπως είπα θα πάει και στη Ρέτζη. Καλό θα ήταν να αναφέρουμε θετικά όλα αυτά τα θέματα. Πολλά μπορούμε να κάνουμε, όλοι οι ευφυείς επιστήμονες που ε, εργάζονται στις περιφέρειες και προσπαθούν να βρουν λύσεις για τα προβλήματα θα πρέπει να είναι σε θέση να αξιοποιήσουν ε, αυτό το μέσο. Όταν ε, συνομιλώ με ανθρώπους από την οικονομία, αυτό που μου λένε είναι ότι θέλουν ευρωπαϊκές προδιαγραφές, ούτω ώστε όταν αναπτύσσουν προϊόντα να είναι συμβατά με τα παρόμοια και με τους τομείς όπως θα χρησιμοποιηθούν, όπου θα χρησιμοποιηθούν σε όλες τις άλλες χώρες. Δεν χρειάζεται να εφευρίσκουμε 100 φορές τον τροχό. Πρέπει να υπάρχει αυτή η συμβατότητα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Όπως είπα υπάρχουν ιδιαίτερα πρικισμένα άτομα σε πολλές εταιρείε που ασχολούνται με αυτά τα θέματα και θέλουν τα προϊόντα τους που έχουν να κάνουν με την παραγωγή και κατανάλωση ενέργειας να είναι ευφυή, να υπάρχει μια ευρία γκάμα πρωτοβουλειών. Για να γίνει αυτό η τυποποίηση είναι ιδιαίτερα σημαντική. Και καταλήγω τονίζοντας ότι ένα πέμπτο των διαθροτικών ταμείων θα χρησιμοποιηθεί για την ε, ε, διανομή της ενέργειας στα πλαίσια του ε, Περιφερειακού Ταμείου, δηλαδή ε, εδώ πρέπει φυσικά να ληφθούν και μέτρα για την ε, αποδοτικότητα της ενέργειας, αλλά αυτές οι εξελίξεις πρέπει να είναι τμήμα και της καινοτομίας για να αντιμετωπίσουμε όλες τις προκλήσεις που έχουμε στο πακέτο ενέργειας. Είναι σημαντικά ποσά αυτά και είχε αναφερθεί το θέμα αυτό και στη Ρέτζη. Πρέπει λοιπόν να επιδιώξουμε να επιτύχουμε τους στόχους μας όπως τους έχουμε περιγράψει στο Horizon 2020, αλλά και περαιτέρω να ε, προσθέσουμε ότι υπάρχουν πολλά πλεονεκτήματα, πολλά ωφέλη από τις νέες τεχνολογίες και θα κερδίσουμε πολλά εάν ε, λάβουμε υπόψη αυτή την πλευρά. Ευχαριστώ και θα υποβάλω πολύ σε αυτή την κατεύθυνση. Υπνά. Ευχαριστώ. Μέχρι στιγμής δεν είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε ορισμένα θέματα που συνδέουν την ενέργεια με τις τεχνολογίες πληροφορικής. Ξέρουμε ότι τα προϊόντα αυτά αναπτύσσονται, αναπτύσσονται πολύ σύντομα, με μεγάλη ταχύτητα. Είναι πρώτη λοιπόν δυνατότητα που έχουμε να συζητήσουμε τέτοια θέματα και ξέρουμε ότι χωρίς καινοτομία, χωρίς έρευνα, δεν θα επιτύχουμε τους στόχους που έχουμε ορίσει. Πρέπει λοιπόν να ε, επικεντρωθούμε σε αυτό που ήδη αναφέρθηκε. Πρέπει να δοθούν οι αναγκαίες πιστώσεις στις περιφέρειες, ε, στην τοπική αυτοδιοίκηση για να αναπτύξουν επί τόπου τεχνολογίες για την ενέργεια αυτές τις λεγόμενες αποκεντρωμένες ε, τεχνολογίες ενέργειας που συμπληρώνουν τα μεγάλα έργα αλλά και αποτελούν και τη σύνδεση ανάμεσα στην παραγωγή ενέργειας και σύγχρονες τεχνολογίες ε, πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Είμαστε στα πρόθυρα μιας ε, κοσμογονικής αλλαγής. Νομίζω ότι φυσικά η παραγωγή ηλεκτρισμού χρειάζεται παντού. Σύντομα θα έχουμε ηλεκτρικά αυτοκίνητα, πολύ περισσότερα και οι περισσότερες από τις οικιακές μας συσκευές θα πρέπει να περιέχουν ε, το αναγκαίο λογισμικό για να ε, κάνουν αποδοτική χρήση της ενέργειας. Θα είναι λοιπόν όλες αυτές οι ηλεκτρικές συσκευές προϊόντα πραγματικά υψηλής και καινοτόμου τεχνολογίας. Πριν λοιπόν αποφασίσουμε πώς θα δαπανίσουμε τα χρήματα, πρέπει να ξέρουμε σε ποια κατεύθυνση θέλουμε να πάμε. Και πιστεύω ότι πρέπει να πάμε στην κατεύθυνση της καινοτομία και της έρευνας. Όχι μόνο για τις ανανεώσιμες. Ορισμένοι τονίσατε τη σημασία των ανανεωσίμων πηγών ενέργειας. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Θα πρέπει να γίνει έρευνα σε όλες τις μορφές ενέργειας που θα μας επιτρέψει ε, να αντιστοιχίσουμε καλύτερα την ζήτηση από τη μία μεριά και άλλες πλευρές από την άλλη. Δηλαδή, να επιτύχουμε τους στόχους μας ε, χωρίς υπερβολικές δαπάνες για τις ε, ε, βιομηχανίες που μπορεί να είναι ιδιαίτερα ενεργοβόρες. Πολλοί Ευρωπαίοι βεβαίως με τρόμο κοιτάζουν τους λογαριασμούς του ηλεκτρισμού Ξέρουμε ότι είναι διπλή, για παράδειγμα, κατά μέσο όρο από τι ΗΠΑ. Άρα, στόχος μας πρέπει να είναι η παραγωγή φτηνής, ταχύτερης, καλύτερη ενέργεια, ε, ε, αξιοποιώντας αξιοποιώντα ε, τι καλύτερε τεχνολογίε, τι καλύτερε συσκευέ. Δεν πρέπει να μα ικανοποιεί η κατάσταση όπου βρισκόμαστε. Πρέπει όντω να προσθέσουμε νέες πλευρές σε αυτό το κείμενο, να επικεντρωθούμε περισσότερο στην ε, καινοτομία στο μέλλον και ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Βιδάλ Ευχαριστώ. Υπάρχουν θέματα πολύ αμφιλεγόμενα στην ενέργεια, τα οποία συχνά συζητούμε και στην Επιτροπή μας και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Αντίθετα λοιπόν με αυτά τα αμφιλεγόμενα ζητήματα, το θέμα των ευφυών ε, δικτύων ε, νομίζω ότι είναι κοινά αποδεκτό και δεν είναι καθόλου αμφιλεγόμενο. Είναι ουσιώδου σημασία ε, τα ευφυή δίκτυα για την καλύτερη μεταφορά και χρήση της ηλεκτρικής ενέργειας και μπορεί να λύσει ε, την παλαίωση των δικτύων, προβλήματα δηλαδή όπως η παλαίωση των δικτύων, η δυσκολία μεταφοράς κτλ. Επομένως πρέπει να καλωσορίσουμε οπωσδήποτε την γνωμοδότηση της συναδέλφου μας Μαρίτα Ουλκουσκόκ ε, η οποία ε, σωστά υπογραμμίζει ότι η σωστή ενσημάτωση ε, της νέας γενιάς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας θα βοηθήσει ε, ε, θα βοηθήσουν μάλλον τα FIA δίκτυα έτσι ώστε να γίνει πιο προσιτή και πιο εύκολη η μεταφορά αυτών των μορφών ενέργειας αυξάνοντας κατά πολύ την ενεργειακή ικανότητα. Επιπροσθέτως να μην λησμονούμε ότι τα FIA δίκτυα θα ωφελήσουν τους καταναλωτές, ε, θα τους δίνουν ακριβείς πληροφορίες για την κατανάλωσή τους. Θα τους δίνουν επίσης την δυνατότητα να παίρνουν καλύτερες αποφάσεις όσον αφορά την κατανάλωση ενέργειας και επομένως να ελέγχουν καλύτερα τον ενεργειακό τους λογαριασμό. Εν παρόδο δεν να πω ότι στην ε, Ισπανία ε, πολύ πρόσφατα είχαμε μια αύξηση κατά 3% του λογαριασμού του ηλεκτρικού. Στην ε, ε, Επιτροπή λοιπόν Περιβάλλοντος που φαίνεται ότι δυσκολεύονται λίγο ε, να δεχτούν το κείμενο στέλνουμε εμείς σαν Επιτροπή Βιομηχανίας ένα πολύ σαφές μήνυμα για το προς τα που θα πρέπει να πάει η ενεργειακή πολιτική τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ και συνάδελφος Χέρτσοκ. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γκριχά. Καταρχάς γνωρίζουμε ότι ο ηλεκτρισμός αυξάνεται, αυξάνεται το ποσοστό του στην ε, χρήση ενέργειας και σε ορισμένα κράτη-μέλη έχει επιβραδυνθεί η κατασκευή ε, εφιών δικτύων και δικτύων γενικότερα. Οπότε η Ρέτζη στην έκθεσή της, στη δική μου έκθεση, και συγχαίρω τη Μαρίτα Ούσκετ που ε, συντάσσει τη γνωμοδότησή μας. Όλοι λοιπόν ε, αναφέρουμε σε αυτή την έκθεση της Ρέτζη ε, γνωρίζουν ότι η αποδοτικότητα της ενέργειας δεν έχει αξιοποιηθεί μέχρι στιγμής πλήρως ούτως ώστε να χορηγούμε αποδοτική ενέργεια στους καταναλωτές είναι η κοιμωμένη του δάσους η αποδοτικότητα. Πολλές δυνατότητες δεν έχουν αξιοποιηθεί. Εάν λοιπόν εγώ στο σπίτι μου κοιτάξω από το παράθυρο της κρεβατοκάμαράς μου βλέπω τους ηλεκτρικούς πυλώνες στους οποίους προστίθενται γραμμές για τη μεταφορά ηλεκτρισμού σε άλλους, ε, σε άλλους πυλώνες προστίθεται γραμμές ε, τηλεφωνίας. Αυτοί οι πυλώνες είναι εκεί από τότε που γεννήθηκα. Και όπως είπε ο Βιδάλ Κουάδρας, στο Πεθρό πολλές φορές ε, τα δίκτυα είναι πολύ μεγάλης ηλικία. Αν θέλουμε να κάνουμε κάτι λοιπόν, αν θέλουμε να υπάρξει πρόοδος, θα πρέπει να αναπτύξουμε μαζί με τα δίκτυα και την, ε, τις τεχνολογίες πληροφορικής και τηλεπικοινωνιών. Γιατί τα ευφυή e δίκτυα ε, πρέπει να συμπεριλάβουν και τον τελικό καταναλωτή. Αυτό όμως έχει και ένα συγκεκριμένο κόστος που πληρώνουν οι καταναλωτές, ιδιαίτερα εάν ε, πρέπει να γίνουν κάποιες επισκευές φέρουν ε, χωριστά ένα μεγάλο τμήμα οι καταναλωτές. Όπως σας είπα, εξετάζουμε το θέμα αυτό και στη Ρέτζη και άμα μελετήσετε την αιτιολογική, την μελέτη επιπτώσεων, θα διαπιστώσετε ότι αναφέρουμε ότι όταν αυξάνουμε το δυναμικό του δικτύου, το 80% ε, αφορά επισκευές και επεκτάσεις. Άρα το θέμα δεν είναι μόνο να αυξήσουμε την αποδοτικότητα, αλλά να αυξήσουμε και την αποδοτικότητα με την οποία δαπανούμε τις πιστώσεις. Διότι ακόμη και στη χώρα μου, αλλά και σε άλλες, δεν έχει αυξηθεί ε, το δυναμικό του δικτύου το τελευταίο διάστημα και πολλές φορές είναι ευάλωτο το ηλεκτρικό δίκτυο για αυτό το λόγο. Θα, πρέπει λοιπόν να υπάρξει συνεργασία μεταξύ των διαφόρων ε, εμπλεκομένων ε, πλευρών και ιδίως για το ευρυζωνικό ίντερνετ. Και εδώ πρέπει να βελτιώσουμε το δυναμικό του συστήματος. Και θα υποβάλω τροπολογίες επ' αυτού. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ, Σέλφος Πρόντι. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και ευχαριστούμε και την Άλφο Ουλσκόγκ για το έγγραφο αυτό το οποίο μας παρουσίασε. Θα ήθελα να αναφερθώ στην σημασία που έχουν τα ΕΦΗ e δίκτυα στην βέλτιστη χρήση των ε, ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Αυτό είναι ιδιαίτερα σημαντικό διότι είναι γεγονός ότι ο κάθε παραγωγός ενέργειας μπορεί να χρησιμοποιήσει τη δικιά του παραγωγή, τη δικιά του ενέργεια κατά προτεραιότητα σε σχέση με την ενέργεια που παρέχεται από το δίκτυο. Υπάρχει και κάτι άλλο σημαντικό. Αυτά τα ευφυή δίκτυα μαζί με μια ε, δυνατότητα μεταφοράς ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στα λεγόμενα super grids μπορούν να βελτιστοποιήσουν την ε, διανομή των ανανεώσιμων ενεργειών που θα πρέπει κατά προτεραιότητα να χρησιμοποιούνται σε σχέση με τις υπόλοιπες μορφές ενέργειας. Επομένως, τα εφή e δίκτυα μαζί με δίκτυα υψηλής αποτελεσματικότητας σε σχέση με τη μεταφορά τους ε, μπορούμε να έχουμε δίκτυα με πολύ μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα, κυρίως δε θα έχουμε δίκτυα ε, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιήσουν στο μέγιστο βαθμό και με το βέλτιστο τρόπο τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας. Κατά αυτήν την έννοια ε, τα εφή δίκτυα θα πρέπει να είναι ευρωπαϊκή προτεραιότητα. Γνωρίζουμε ότι οι εθνικοί οργανισμοί θα αντιταχθούν αλλά θα πρέπει να ξεπεραστεί το πρόσκομα αυτό γιατί ε, όλοι θα ωφεληθούμε από την ε, λειτουργία των ευφυών δικτύων. Ευχαριστώ πολύ. Συνάδελφε πρώτη η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Thank you, Madam Ευχαριστώ και καλημέρα. Φαν ναι, εκλέγομαι και είμαι επικεφαλής ε, τμήματος ε, και γενικός της Γενικής Διεύθυνσης ε, Ενέργειας. Ασχολούμαι με την ηλεκτρική ενέργεια. Ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να σχολιάσω την έκθεση. Προέκυψε με σαφήνεια νομίζω από τη συζήτηση ότι στη γνωμοδότηση υπάρχουν εύστοχα στοιχεία για τα ευφύ δίκτυα και χαιρόμαστε που είναι τόσο ευρία η συνένεση με το Κοινοβούλιο σε σχέση με το τι πρέπει να γίνει. Δεν χρειάζεται να αναφερθώ σε όλα τα σημεία. Συνέργεια με τις νέες τεχνολογίες, με τα δυνατότητα μεταφοράς, νέες δυνατότητες διανομής και το καθεξής. Είναι σημαντικό να αναφερθούμε όχι μόνο στη σημασία για τους καταναλωτές, αλλά και το πολύ σημαντικό θέμα της προστασίας ε, των δεδομένων. Πέραν αυτού του ζητήματος πρέπει να μιλάμε και για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των καταναλωτών αυτής καθ' αυτής. Επίσης ε, ζητάτε μια νέα διατύπωση για να τονιστεί ο ρόλος ε, και η σημασία των τοπικών πρωτοβουλίων και των ε, προγραμμάτων περιφερειακής ανάπτυξης. Αυτό προσπαθούμε και εμείς και επιδιώκουμε να ενσωματώσουμε στο κείμενο για τις τοπικές πρωτοβουλίες. Θα ήθελα να τονίσω ότι δεν περιοριζόμαστε στις πολυάριθμες τέτοιες πρωτοβουλίες σε εθνικό επίπεδο αλλά και σε ευρωπαϊκές πρωτοβουλίες όπως ε, ε, οι πρωτοβουλίες του Σώματος των Δημάρχων ε, και προωθούμε αυτή την πρωτοβουλία με το που δρομολογήθηκε η ετήσια τελετή γίνεται στην Ολομέλεια, στην αίθουσα της Ολομέλειας του Κοινοβουλίου ετησίως και καλό θα ήταν σε αυτή την ε, συντακτική συνέλευση των δημάρχων ε, να αναφερθούμε συγκεκριμένα στα ΕΦΗ δίκτυα φέτος. Επίσης, ε, τονίζεται η σημασία των προτύπων αυτό συνδυάζεται με την έμφαση που δίνουμε στις περιφερειακές δράσεις, γιατί οι δράσεις θα πρέπει να γίνονται στο κατώτερο δυνατό επίπεδο, ε, όσο το δυνατόν εγκύτερα γίνεται ε, στον καταναλωτή. Συνεργαζόμαστε και με τους οργανισμούς τυποποίησης αρκετά στενά, αλλά ε, φυσικά θα αξιοποιήσουμε οποιαδήποτε επιπλέον πλέον ε, όθηση μας δώσει το Κοινοβούλιο. Τελευταία παρατήρηση. Αν υπάρχει ε, κάτι που λείπει κατά τη γνώμη μας από τη γνωμοδότηση και δεν ακούστηκε και στη σημερινή συζήτηση όμως εμείς κρίνουμε ότι αξίζει να ε, τονιστεί είναι η διασύνδεση ανάμεσα στα ευφυή δίκτυα και την εσωτερική αγορά. Πρέπει να ξεκαθαριστεί ότι ο στόχος δεν είναι να προσφέρουμε ωφέλη στους καταναλωτές σε περίπτωση που δεν ολοκληρωθεί η εσωτερική, ενέργεια ηλεκτρικής, ε, εσωτερική συγγνώμη, αγορά ηλεκτρικής ενέργειας είναι αναπόσπαστο κομμάτι, είναι ένα εργαλείο που θα μας βοηθήσει για να ολοκληρώσουμε την ε, εσωτερική αγορά της ηλεκτρικής ενέργειας και είναι νομίζω σημαντικό να ε, τονίσουμε και αυτή την πτυχή. Επίσης μιλήσαμε για τα ωφέλη προς τους καταναλωτές μέσω της περαιτέρω ανάπτυξης της ενιαίας εσωτερικής αγοράς ηλεκτρικής ενέργειας, τα FEE e δίκτυα θα είναι ένας από τους τρόπους που θα επιτευχθεί αυτό και θα είναι υποφελής για τους καταναλωτές. Στο σημείο λέμε ότι δεν πρέπει να φέρουν το οικονομικό βάρος ε, οι καταναλωτές, ε, πολύ εύστοχο και αξίζει να το υποστηρίξουμε, αλλά ας μιλάμε για το καθαρό οικονομικό βάρος, γιατί τα εφή δίκτυα απαιτούν σοβαρές επενδύσεις, όμως είναι σημαντικό να μην υιοθετηθούν οι φθηνότερε λύσεις μόνο και μόνο για να εξοικονομηθούν κονδυλία. Είναι σημαντικό όταν επενδύσουμε να ξεκαθαρίσουμε και ποια είναι τα καθαρά ωφέλη που τελικά θα καρποθούν οι καταναλωτές. Και συχνά ε, ε, συμβαίνει το εξή ότι όσο υψηλότερε είναι επενδύσει, τόσο μεγαλύτερα είναι τα ωφέλη στη συνέχεια. Και θα σταματήσω εδώ. Ευχαριστούμε. Θα ακούσουμε τώρα την συνάδελφο Ουλφσκοκ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε και θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για όλες τις παρεμβάσεις τους. Όπως είπε η συνάδελφος Χέρτσοκ, είναι κάτι το απαραίτητο ε, όμως ακόμη είναι σε ένα λίθαργο αυτό το πρόγραμμα των υφείων δικτύων, δεν έχει πλήρως αναπτυχθεί. Και όπως είπε ο κύριος Βιτάλ Κουάντρας, δεν είναι αμφιλεγόμενο αυτό το ζήτημα. Όλοι συμφωνούμε και υπάρχει ομοθυμία ακόμη και με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, όχι μόνο στις πολιτικές ομάδες του Κοινοβουλίου. Ταυτόχρονα ξέρουμε ότι ε, τη της οικονομικής κρίσης μειώθηκαν στο ελάχιστο οι επενδύσεις σε όλους τους τομείς, ακόμη και ε, σε τομέα που χρειάζονται ε, τόσο πολύ όπως τον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Ε, έχουμε λοιπόν το 1 πέμπτο των κονδυλίων των διαρθρωτικών ταμείων που διοχετεύονται σε αυτό το τομέα της ενέργειας. Ταυτόχρονα θα έπρεπε να βρούμε και άλλες πηγές ε, χρηματοδότησης, ε, διότι δεν πρόκειται μόνο για περιφερειακή ανάπτυξη. Σχετίζεται αυτό με την έρευνα και την ανάπτυξη και ως εκ τούτου θα έπρεπε να διαφοροποιήσουμε τις πηγές χρηματοδότησης και αυτό το λέω εν ώψη των μελλοντικών βημάτων που θα κάνουμε για να γίνει ευρύτερη χρήση αυτής της νέας τεχνολογίας. Τώρα, ε, το πώς θα χρησιμοποιηθούν ε, τα διάφορα είδη κονδυλίων και γραμμών προϋπολογισμού στον τομέα της ενέργειας, ε, θα έλεγα ότι για να προωθήσουμε τις επενδύσεις ε, στα FEE δίκτυα θα πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο διασυνδεμένο είναι το ζήτημα με άλλα βασικά ζητήματα της πολιτικής Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, εξάλλου είναι και πολύ μακρύς ο χρονικός ορίζοντας, ε, σχεδόν 50 χρόνια. Ε, η συνάδελφό ε, Χίμπνερ, ε, Νίστελ Ρόι, Βίτελ Πρόντι και Χέρτσοκ όλοι τόνισαν πόσο σημαντικό είναι το ζήτημα για θέματα έρευνας και κοινοτομία. Ε, τώρα, το θέμα της προστασίας των δεδομένων. Είναι ξεκάθαρο ότι είναι ιδιαίτερα επίκαιρο αυτό το ζήτημα τώρα για άλλους λόγους. λόγω των κλειδονισμών που προκάλεσαν οι ελλείψεις που διαπιστώθηκαν στο σύστημα προστασίας ε, των προσωπικών δομένων και της προσωπικής ε, ακαιρεότητα. Εξυπακούεται ότι με ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να το ζήτημα, κυρίως τα ευφυή e e δίκτυα που μετρούν την καθημερινή μας δραστηριότητα μέσα στα σπίτια μας. Ε, και έτσι θα εξασφαλίσουμε ε, ωφέλη για τους καταναλωτές με ασφάλεια όμως. Ε, τα ωφέλη των καταναλωτών ε, συνδυάζονται με τα ωφέλη που θα έχουμε από τα σπίνος, δηλαδή παράγωγα προϊόντα ή επενδύσεις που θα διοχετευτούν σε άλλους τομείς εάν επιτευχθούν ε, στον τομέα της ηλεκτρικής ενέργειας. Δεν περιοριζόμαστε στα εφηδίκτυα. δίκτυα. Λοιπόν, για να κλείσω, να σας ευχαριστήσω και πάλι. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το ζήτημα και επανειλημμένα και σε διάφορα βήματα το έχουμε συζητήσει ε, τα τελευταία χρόνια, κυρίως κατά την τωρινή θητεία και στα πλαίσια των εργασιών της Επιτροπής μας, μας έχει απασχολήσει επανειλημμένα το ζήτημα ε, και θα καταβάλω κάθε δυνατή προσπάθεια του ώστε να συμπεριλάβω όλα τα σχόλια που κάνατε σήμερα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ τη συνάδελφο. Την ε, Παρασκευή 4 ε, Νοεμβρίου λίγη προθεσμία για την υποβολή τροπολογιών. Ε, θα σταματήσουμε μέχρι τις 10, γιατί στις 10 θα ξεκινήσει η ηλεκτρονική ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Bene, Καθίστε σας παρακαλώ. Έχουμε σημαντικές και πολλές ψηφοφορίες. Επομένως, να καθίσετε έτσι ώστε να κάνουμε πρώτα έναν έλεγχο για την ηλεκτρονική ψηφοφορία και μετά να ξεκινήσουμε. να κάνουμε λοιπόν πρώτα έναν έλεγχο. Έχετε τις κάρτες ψηφοφορίας. Βάλτε λοιπόν στη θέση της την κάρτα για να κάνουμε έναν έλεγχο. Ψηφίστε. Aujourd'hui, si y a un peu pas, je ne prends parce que je dois voter. Votazione chiusa. Πέρα τη ψηφοφορία. Πολύ ωραία. Έχουμε 28. Α, όχι, όχι, κάποιοι δεν είχαν ψηφίσει. Να ξανανοίξουμε λίγο, να ξαναξεκινήσει η ψηφοφορία για τελευταία φορά έλεγχος. Ψηφίστε ναι. Α, ο κύριος Πρώτη δεν είχε ψηφίσει. Απόστο τούτη, πληροφορια κιούζα. Πέρας της ψηφοφορίας. ...37 παρόντες συν ο συνάδελφος πρώτη που ξέχασε την κάρτα του. Λοιπόν, πριν ξεκινήσουμε την ψηφοφορία, γιατί μετά δεν θα καταφέρω να το κάνω, να σας πω το εξής. Στο τέλος της ψηφοφορίας, παρακαλώ πολύ τους συναδέλφους και όλους τους άλλους παριστάμενους να εγκαταλείψουν την αίθουσα με ταχύτητα, γιατί κάθε φορά μετά το πέρας της ψηφοφορίας χάνουμε 7-8 λεπτά περιμένοντας να φύγουν όσοι δεν ενδιαφέρονται για τη συνέχεια από την αίθουσα. Λοιπόν, δύο λεπτάκια. Όσοι θέλουν να φύγουν, να φύγουν. Όσοι θέλουν να μείνουν, να μείνουν στην αίθουσα. Επίσης, ε, πριν ξεκινήσουμε την ε, ψηφοφορία για το Horizon, η συνάδελφος ε, Χέμπνερ ζήτησε αν είναι δυνατόν να ψηφιστεί η δικιά της έκθεση, που είναι μια ενιαία ψηφοφορία γιατί έχει μια υποχρέωση και πρέπει να φύγει. Ξεκινάμε λοιπόν με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Θα ψηφίσουμε την έκθεση της συναδέλφου Ήπνερ είναι το σημείο 25. Είναι μία και μόνη ψηφοφορία. Η έκθεση της κυρίας Χίμπνερ, διάσκεψη Ηνωμένων Εθνών για την αλλαγή του κλίματος. Γιολάντα Εμιλία Ήμπνερ, ΚΟΠ 19 για την κλιματική αλλαγή. Το βρήκατε, είναι το σημείο 25 της μερικής διατάξεως. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 37 ψήφοι υπέρ, 5, 38 ψήφοι υπέρ, 5 κατά, καμία ε, αποχή Συγχαρητήρια συνάδελφε Χίπνερ. Έκθεση Κρότσμαν. Που αφορά το κόσμο, παρακαλώ. Εκπροσωπώ τον κύριο Κρότσμαν. Θέλει να κάνει μία δήλωση για να γίνει κατανοητό, γιατί δεν είναι σαφή τα στοιχεία, τα νούμερα. Η δήλωση του εισηγητή για τον τριμερή διάλογο για το κόσμο πριν ψηφίσουμε το κείμενο του συμβασμού, ο κύριος Κρόισμαν θέλει να μπει στα πρακτικά ότι το κείμενο χρειάζεται ακόμη μερικές τεχνικές προσαρμογές πριν περάσει για ψηφοφορία στην Ολομέλεια. Τα αριθμητικά στοιχεία για το συνολικό προϋπολογισμό έχουν εκφραστεί με σταθερές τιμές, αλλά για να είναι σωστά πρέπει να μεταφραστούν στις ε, σημερινές τιμές για να λάβουν υπόψη τον πληθωρισμό τα επόμενα 7 χρόνια το ποσό για τα χρηματοδοτικά μέσα δεν θα πρέπει να είναι απόλυτα στοιχεία, αλλά ως ποσοστό περίπου 60% δηλαδή του προπολογισμού. Πρόκειται για μια καθαρά τεχνική προσαρμογή, διότι τα τρία θεσμικά όργανα συμφωνούν για τα θέματα αυτά και ανταποκρίνονται στην συνήθη διαδικασία. Η Γραμματεία πριν την ψηφοφορία στην Ολομέλη θα κάνει τι αναγκαίε προσαρμογές στο κείμενο. Ευχαριστώ πολύ. Πολύ ωραία. Με αυτή την αποσαφήνιση ψηφίζουμε την έκθεση Κρόιτσμαν. Άρχεται η ψηφοφορία. Votazione chiusa. Πέρα της ψηφοφορίας. Έχουμε μία ψήφο ΕΛΚ ε, πλεονάζουσα. Ωραία βγάλατε την κάρτα σας. 44 υπέρ, 2 κατά, μία αποχή. Εγκρίνεται. Υπολογίζω και τον κύριο Πρόντι που δεν έχει την κάρτα του. Έκθεση Μαντουρέλ. Ψηφίζουμε την έκθεση της κυρίας Μαντουρέλ, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 46 ψήφοι υπέρ, καμία αποχή, καμία ψήφος κατά, εγκρίνεται. Ψηφίζουμε επί της εκθέσεως Καρβάλιο. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 48 υπέρ, καμία αποχή, καμία ψήφος κατά εγκρίνεται. Έκθεση Έλερ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 43 ψήφοι υπέρ, 2 ψήφοι κατά, 1 αποχή εγκρίνεται. Έκθεση Λάμπερτς. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 46 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή, επομένως εγκρίνεται. συνάδελφος Ματίας ε, ζητά συγγνώμη, δεν, είναι, δεν μπορεί να είναι παρούσα, παρόλα αυτά εμείς ψηφίζουμε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 46 ψήφοι υπέρ, 3 κατά, καμία αποχή. Εγκρίνεται η έκθεση Ματίας. Έκθεση Κρόιτσμαν. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Έχουμε ένα, μία ψήφο ΕΛΚ παραπάνω. Ξαναρχίζει η ψηφοφορία, έγινε και ένα λάθος. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. Λοιπόν, 20 ψήφοι υπέρ, 24 ψήφοι κατά, 3 αποχές, επομένως απορρίπτεται. Περνάμε στην έκθεση Τροτμάν. Τροπολογία 39 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 41 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 43 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47 και τροπολογία 48 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 και 51 μαζί υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 52 υπέρ κατά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 71 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 72 μαζί με την 73 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 74 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 76 και 77 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. 75 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 83 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90 υπέρ 90 ναι, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 4 ίγκο υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 15 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 85 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται Έλεγχος ηλεκτρονικός για την τροπολογία 85, μάλιστα. Πέρας. 23 υπέρ, 24 κατά απορρίπτεται. Μάλλον 25 κατά. Απερίφθη. 86 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 87 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 88 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 89 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ψηφίζουμε on αφού υπάρχει συμφωνία όλες τις τροπολογίες ΥΜΚΟ 1 έως 16 υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 91 υπέρ κατά αποχέ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 κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 13, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 14, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογίες 15, 16 και 21, υπέρ κατά αποχές εγκρίνονται, τροπολογία 17 μαζί με την 29 προφορική τροπολογία, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, τροπολογία 18, υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογίες 19 και 20 μαζί, υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνονται. Τροπολογία 24. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 25 μαζί με την 38. Υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 μαζί με την 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 26 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογίες 31 και 32 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονικός έλεγχος για τις τροπολογίες 31 και 32. Δήμαρχος για τις τροπολογίες 31 και 32. Έχει ψηφίσει ένας Ελκ Παραπανίσιος και ένας από τους ε, σοσιαλιστές και δημοκράτες. ΕΛΚ λοιπόν και οι σοσιαλιστές ε, πρέπει να διορθώσουν την ψήφο. Πολύ ωραία, πέρας της ψηφοφορίας. Πέρας της ψηφοφορίας. 24 ψήφοι υπέρ, 25 ψήφοι κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 33. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 34. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 35. Υπέρ. Με προφορική τροπολογία πρέπει να σας το πω. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. Τροπολογία 36. Υπέρ. Κατά. Εγκρίνεται. 37. Υπέρ κατά εγκρίνεται τελική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Έχουμε εν, μία ψήφο παραπάνω από τους σοσιαλιστές, διορθώθηκε το λάθος αυτό, ωραία. Ψήφι 50 υπέρ συγχαρητήρια. Περνάμε στην έκθεση Βαλεάν. Συμβιβασμός 2 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 37 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 3 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 38 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 40 Α, τροπολογία 39, υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 40, υπέρ. Κατά αποχές να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας, έχουμε μία ψήφο παραπανίσια. Πέρας. 23 ψήφοι υπέρ, 26 κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 41 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 45 υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 46 υπέρ, κατά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 κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 53 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 54 και 44 μαζί υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 55 Θέλετε έλεγχο για τις τροπολογίες 54 και 44 που ψηφίστηκαν από κοινού. Παρακαλώ. Πέρας. Ε, μία ψήφος έλκ παραπανήσια. 28 υπέρ, 22 κατά εγκρίνονται. Ζητώ συγγνώμη. Τροπολογία 55 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 11 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 56, 57 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 58 υπέρ έχει εκπέσει 58. Είχαμε εγκρίνει την τροπολογία 11. Η 56 λοιπόν έχει καταπέσει. Ναι, εγκρίναμε μετά την 57 και τώρα την 58. Πρέπει να ψηφίσουμε την τροπολογία 58. Θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο για την τροπολογία 57. Άρχεται η ψηφοφορία επί της τροπολογίας 57. Πέρας. Ψήφι 21 υπέρ, 28 κατά, απορρίπτεται. Ψηφίζουμε την τροπολογία 58 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Το 12, τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 59 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 61 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 61, παρακαλώ. Τροπολογία 61. Ηλεκτρονική επαλήθευση πέρας της ψηφοφορίας. 25 ψηφί, υπέρ, 25 κατά, επομένως απορρίπτεται. Τροπολογία 62 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Έλεγχος για την τροπολογία 62 παρακαλώ. Πέρας της ψηφοφορίας. Α, Ζητώ πραγματικά συγγνώμη. 37 ψήφοι υπέρ, 12 κατά εγκρίθηκε. Τροπολογία 15 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 67 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. 65 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται 66 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 71 71 μόνη της υπέρ κατά αποχές η ηλεκτρονική επαλήθευση δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα τροπολογία 71 άρχεται η ψηφοφορία πέρας 24 ψήφοι υπέρ, 23 κατά, επομένως εγκρίνεται. Περνάμε τώρα στην τροπολογία 75 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 76 υπέρ, κατά, αποχές ε, είναι ίσα ίσα το αποτέλεσμα Επομένως ψηφίζουμε 76 και 77 μαζί γιατί είναι ταυτόσιμες. Πέρας της ψηφοφορίας, μία ψήφος ΕΛΚ και μία ψήφος σοσιαλιστών πλεονάζουσα. Εντάξει. Έχουμε μία ψήφο σοσιαλιστών παραπάνω εντάξει με το ΕΛΚ, εντάξει με τους σοσιαλιστές. Λοιπόν, πέρα στις ψηφοφορίες, 34 ψήφοι υπέρ, 15 κατά, επομένως ε, εγκρίνονται. 78 και 43 τώρα ψηφίζουμε μαζί, υπέρ, κατά, αποχές, ε, απορρίπτονται. Τροπολογία 19, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 79, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 80 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 20 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 22 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 23 υπέρ κατά απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 23 άρχεται. Πέρας της ψηφοφορίας. 24 ψήφοι υπέρ, 26 κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 24 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 25 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται Συμβασμός 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 3 με προφορική τροπολογία υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 28 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 31 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται και η τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία επί των τροπολογιών. Ε, μία ψήφος ΕΛΚ παραπάνω πέρας της ψηφοφορίας. Εξακολουθεί να υπάρχει μία ψήφος παραπάνω από το ΕΛΚ. Ωραία, πέρα της ψηφοφορίας, 43 ψήφοι υπέρ, 3 αποχές, 3 ψήφοι κατά. Ε, περνάμε στην ε, στη ψηφοφορία τώρα, πάλι με ηλεκτρονική ψηφοφορία, νομοθετικό ψήφισμα. Votazione chiusa. ψηφοφορία. 44 ψήφοι υπέρ, 3 ψήφοι κατά, 3 αποχές. Τελική, μία ακόμα τελική ψηφοφορία όσον αφορά την, την θεσμική διαπραγμάτευση. Ε, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 49 ψήφοι υπέρ, καμία αποχή, καμία ψήφος κατά. Πάρα πολύ ωραία. Συγχαρητήρια. Ολοκληρώσαμε Περνάμε τώρα στην έκθεση της ε, συναδέλφου Τόια. Τροπολογία 38. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 39. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. Τροπολογία 40. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 41 και 42 από κοινού είναι ταυτόσιμες υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Αν θέλετε ηλεκτρονικό έλεγχο, ναι, ναι, βεβαίως, να κάνουμε ηλεκτρονικό έλεγχο, 41-42. 41-42 μαζί. Πέρας. 27 ψήφοι υπέρ, 21 ψήφοι κατά, επομένως εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 12 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 44 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 45 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 46 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 47 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 49 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 50 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονικός έλεγχος για την τροπολογία 50. Πέρας της ψηφοφορίας. 8 ψήφοι υπέρ 40 κατά, επομένως απορρίπτεται. Τροπολογία 14. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 51. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 52. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. 15. Υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. 54. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Ε, ηλεκτρονική επαλήθωση για το 54. Α, ναι, ναι, έκανα λάθος. Έκανα λάθος, έχετε δίκιο. Εν πάση περιπτώσει. Πέρας της ψηφοφορίας. Ε, ναι, βεβαίως. Ε, ε, έχει... Ε, είναι κατά η ψηφοφορία. η 55 υπέρ κατά αποχές τι να σας πω. Δεν ξέρω. 55, 55 ηλεκτρονική επαλήθευση. Πέρας. 27 27ψηφί υπέρ, 21 21ψηφί κατά, επομένως εγκρίνεται. 56. Κατά. Εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά εγκρίνεται. 58 υπέρ κατά εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ηλεκτρονική επαλήθευση επί του 58. 58. Ε, ηλεκτρονική ψηφοφορία επί της τροπολογίας 58 πέρας. 19 ψήφοι υπέρ, 27 κατά, επομένως απερίφθη. Η 59 έχει εκπέσει από ό,τι μου λένε και γι' αυτό ψηφίζαμε την τροπολογία 58 διότι είχαμε απορρίψει την τροπολογία 54. Γι' αυτό δεν ψηφίσαμε την τροπολογία 59 και μόλις ψηφίσαμε την τροπολογία 58. ...58, λοιπόν η οποία απερίφθη. Ψηφίζουμε από κοινού τις τροπολογίες 60, 61 και 62 μαζί. Υπέρ, κατά, Αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Ε, ψηφίζουμε για τις τροπολογίες 60, 61 και 62. Πέρας της ψηφοφορίας απερίφθη. Τροπολογία 16. Υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 63. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 63. Πολύ ωραία. Πέρας. 24 ψήφοι υπέρ, 25 κατά απερίφθη. Τροπολογία 17. Υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 64. Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 65. Υπέρ κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 66 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 67 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 68 υπέρ. Κατά. Αποχές. Προτιμώ να κάνουμε επαλήθευση. Άρχεται η ψηφοφορία. Επί της τροπολογίας 68 πέρας. 30 ψήφοι υπέρ, 20 κατά, επομένως εγκρίνεται. Τροπολογία 69 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 70 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 71 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 72 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 18 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 73 υπέρ. Κατά. Δεν είναι σαφές το αποτέλεσμα. Ηλεκτρονική ψηφοφορία λοιπόν για την 73. Πέρας της ψηφοφορίας Απερίφθη. 74 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 75 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 76 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 77 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 78 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 79 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 79. Παρακαλώ, ψηφίσετε. Έχουμε έναν σοσιαλιστή παραπανίσιο. Τώρα είμαστε εντάξει. 7 ψήφοι υπέρ, 43 κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 80. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Απορρίπτεται. 81. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 83. Υπέρ. Κατά. Αποχές. Εγκρίνεται. Τροπολογία 19. Υπέρ κατά, αποχές απορρίπτεται. 84 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 20 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 85 υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 86 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 86. Πέρας. 32 ψήφοι υπέρ, 18 κατά, επομένως εγκρίνεται η τροπολογία 86, 87 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται 88 υπέρ, κατά. Αποχές απορρίπτεται 89 υπέρ, κατά. Αποχές εγκρίνεται 90, 92 διορθώνει η πρόεδρος υπέρ, κατά αποχές απορρίπτεται. 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 90 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 94 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 95 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 96 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 97 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 98 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 99 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 100 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 101 υπέρ κατά αποχές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 αποχές απορρίπτεται. 29 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 3 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 4 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 30 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 30 ένα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 32 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 33, 34 και 35 από κοινού υπέρ τροπολογία 33 και τις τρεις τροπολογίες μαζί, τροπολογίες 33, 34 και 3 από κοινού. Υπέρ. Κατά. Ηλεκτρονική επαλήθευση. Τροπολογίες 33, 34 και 35. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 20 ψήφοι υπέρ 30 κατά, επομένως απορρίπτονται. Τροπολογία 8 υπέρ κατά. Αποχές να κάνουμε ηλεκτρονική επαλήθευση για την τροπολογία 8 παρακαλώ. Πέρας. 23 ψήφοι υπέρ, 28 κατά, επομένως απορρίπτεται. Τροπολογία 9 υπέρ κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 10, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 11, υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. 36, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 37, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Ε, άρχεται η ψηφοφορία, τελική ψήφος. Πέρας. Έχουμε μία ψήφο σοσιαλιστών παραπάνω. Μία παραπανήσια ψήφος λοιπόν από τους σοσιαλιστές. Πέρας της ψηφοφορίας. 37 ψήφοι υπέρ, 14 ψήφοι κατά, συγχαρητήρια στην εισηγήτρια, διότι εγκρίθηκε η έκθεσή της. Περνάμε τώρα στην έκθεση Τζαβέλα. Τροπολογία 44 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 45 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 47 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 49 υπέρ. Κατά. Αποχές απορρίπτεται. 50 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 51 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 52 υπέρ 52 52 τροπολογία 52 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 55 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Συμβιβασμός 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 63 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 64 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 7 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 78 υπέρ 68 συγγνώμη, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 69 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 70 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 71 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται, 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται, 72 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 73 ε, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβιβασμός 8 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 79 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 82 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 83-85 από κοινού υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 86 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται συμβιβασμός 9 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 90 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 91 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται τροπολογία 92 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 93 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 90, συγγνώμη συμβιβασμός 10 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται τροπολογία 101 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται ε, η ηλεκτρονική επαλήθευση επί της τροπολογίας 101. Άρχεται η ψηφοφορία. Επί της τροπολογίας 101. Πέρας. 21 ψήφοι υπέρ, 23 ψήφοι κατά απορρίπτεται. Τροπολογία 102 υπέρ. Κατά αποχές απορρίπτεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση από τις τροπολογίες 102 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας της ψηφοφορίας. 22 ε, υπέρ, 24 ψήφι κατά, απορρίπτεται. Τροπολογία 103. Υπέρ. Κατά. Αποχές ε, εγκρίνεται. Τροπολογία 12. Υπέρ, κατά, αποχές ε, εγκρίνεται 104 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται 105 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 106 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 107 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 108 Α, θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση από τις τροπολογίες 107. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας. 21 ψήφοι υπέρ, 26 κατά, επομένω απορρίπτεται. 107, τροπολογία 107 απερίφθη. Τροπολογία 108 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 109 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 110 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 111 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. 113 υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Ηλεκτρονική επαλήθευση από τις τροπολογίες 113. Πέρας της ψηφοφορίας. 24 ψήφοι υπέρ, 23 ψήφοι κατά, επομένως εγκρίνεται. Τροπολογία 114. Άρχι... Υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 115 υπέρ. Κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 116 υπέρ. Τι θέλετε, η ηλεκτρονική επαλήθευση επί της 115. Πολύ ωραία. Τροπολογία 115, ηλεκτρονική ψηφοφορία, άρχεται η ψηφοφορία. Πέρας η ψήφη είναι 36 υπέρ 10 κατά, επομένω εγκρίνεται. 116 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 117 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 118 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Από κοινού 119, 120, 121 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 13 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 122 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 123 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 124 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. 125 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 126 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 14 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 127 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση από τις τροπολογίες 127 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. 23 ψήφοι υπέρ, 24 κατά, απερίφθη. Τροπολογία 14. Τροπολογία 14. Υπέρ, κατά, αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 15. Υπέρ, κατά, αποχές απορρίπτεται. 128. Υπέρ, κατά, απορρίπτεται. 129 και 130 μαζί, υπέρ, κατά εγκρίνεται. 132 υπέρ κατά Νομίζω ότι απορρίπτεται, αλλά καλύτερα να το επαληθεύσουμε. Η ηλεκτρονική επαλήθευση από τις τροπολογίες 132. 132, πέρας της ψηφοφορίας. 41 ψήφοι υπέρ, 2 κατά, εγκρίνεται. 133 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. 135 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 136 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 137 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 138 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 139 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 16 υπέρ. Κατά. Απερίφθη τροπολογία του κ. Ζαντό. Η τροπολογία 17 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 18 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 19 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 19 παρακαλώ. Άρχεται η ψηφοφορία. Πέρα τη ψηφοφορία. 23 ψήφοι υπέρ, 21 κατά εγκρίνεται. Τροπολογία 20 υπέρ, κατά. απόχέ απορρίπτεται. Συμβιβασμό 1 υπέρ, κατά. απόχέ εγκρίνεται. Τροπολογία 21 υπέρ, κατά. απόχέ απορρίπτεται. Τροπολογία 22, όχι. Α, τροπολογία 1. Πηγαίνουμε στην τροπολογία 1, υπέρ. Κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 24, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 25, υπέρ. Κατά, αποχές, απορρίπτεται. 26, υπέρ. Κατά, αποχές απορρίπτεται. Τροπολογία 27 πρώτο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 27 δεύτερο τμήμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 28 υπέρ κατά αποχές ηλεκτρονική επαλήθευση της τροπολογίας 28. Πέρας. 21 ψήφοι υπέρ, 26 κατά, επομένως απερίφθη τροπολογία 28. Τροπολογία 2 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Συμβιβασμός 3 υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Τροπολογία 36 υπέρ, κατά, αποχές, απορρίπτεται. Τροπολογία 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται, συμβιβασμός 4 υπέρ, κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 5 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 6 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 40 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 41 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 42 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Τροπολογία 43 υπέρ κατά αποχές απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία. Θέλετε ηλεκτρονική επαλήθευση από τη τροπολογία 43. Παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Τροπολογία 43, ηλεκτρονική ψηφοφορία. Πέρας. 23 ψήφοι υπέρ, 24 ψήφοι κατά, απορρίπτεται. Τελική ψηφοφορία με ηλεκτρονική ψηφοφορία. Παρακαλώ πέρα της ψηφοφορίας. Και τώρα έχουμε την έκθεση Δεν σας είχα πει το αποτέλεσμα για την προηγούμενη ψηφοφορία. 42 υπέρ, 2 ψήφοι κατά, 1 αποχή. Εγκρίνεται λοιπόν και συγχαίρουμε την εισηγήτρια. Περνάμε τώρα στην έκθεση Beauty Coffer. Μία ηλεκτρονική ψηφοφορία. Άρχεται. Συνάδελφε Έλερ. Απλώς... Λόγους ε, πρακτικών. Ψηφίσαμε την πρόταση για το Horizon 2020. Καμία από τις πρωτοβουλίες ε, του Κοινοβουλίου δεν αναφέρεται στον προπολισμό του Συμβουλίου. Δεν πρέπει να σταματήσει εδώ αυτή η διαδικασία στην Ήτρε. Πρέπει να έχουμε υπόψη μας ότι το Συμβούλιο δεν συμπεριέλαβε καθόλου τις πρωτοβουλίες μας ε, στον προπολογισμό και σε διαβούλευση με τα άλλα θεσμικά όργανα κατά την ψηφοφορία στην Ολομέλεια πρέπει να συμπεριληφθεί. Γιατί αλλιώ ό,τι κάναμε τα τελευταία δυόμιση χρόνια γελιοποιείται. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ, πολύ συνάδελφε Τελική ψηφοφορία επί της εκθέσεως Μπουτικόφερ άρχεται. πέρας της ψηφοφορίας. 42 ψήφοι υπέρ, καμία ψήφος κατά, τέσσερις αποχές. Εγκρίνεται λοιπόν και συγχαίρουμε τον συνάδελφο Μπουτικόφερ. Και αυτό ήταν το τέλος της ώρας των ψηφοφοριών. Ε, κάναμε όλες τις ψηφοφορίες που είχαμε γράψει στη μερίσια διάταξη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ε, δύο-τρία λεπτάκια έτσι ώστε να φύγουν ε, όσοι δεν θέλουν να παραμείνουν στην αίθουσα και να προετοιμάζεται ο συνάδελφος Οντή.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 c'est mieux de l'attendre ou non Non, non, non, vous commencez. Dando subito la parola al collega Odi. Eh, να δώσω το λόγο στον συνάδελφο Οντή για να μας παρουσιάσει την έκθεσή του για την τεχνολογική βάση της Ευρωπαϊκής Αμυντικής Βιομηχανίας. Έχουμε περιορισμένο χρόνο. Βέβαια, ε, σήμερα το πρωί, αλλά παρακαλώ έχετε το λόγο. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Υπενθυμίζω σύντομα το πλαίσιο. Ο πρόεδρος Φαν αποφάσισε να υπάρξει έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στα μέσα Δεκεμβρίου για να συζητήσει με τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων για τις, τους προσανατολισμούς ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης για θέματα ασφάλειας και άμυνας και γι' αυτό η Υποεπιτροπή για την Άμυνα και η ΑΦΕΤ ξεκίνησαν μια συζήτηση, ευχαριστώ πολύ. Ε, όπως σας είπα και προηγουμένως αποδέχτηκαν η Επιτροπή μας βάσει το άρθρο 50 να συνεργαστεί για τις βιομηχανικές πλευρές του θέματος. Η γνωμοδότησή μας λοιπόν ασχολείται κυρίως με την βιομηχανική πλευρά, έρευνα, και σε μικρότερο βαθμό ενέργεια. Ήδη κάνουμε μια ανταλλαγή απόψεων. Τώρα εξετάζουμε τις τροπολογίες. Υπήρξαν ε, κάτι λιγότερο από 100 τροπολογίες. Ευχαριστώ τους εισηγητές των ε, άλλων ομάδων τον κύριο, τον κύριο τον κύριο Σανάφσκι, την Ντίνα Ιωάννα Βαλεάν που παρακολούσαν το θέμα αυτό. Τους συνάντησα όλους, συνάντησα και όλους, ευχαριστώ μάλλον και τους άλλους συναδέλφους που υπέβαλαν τροπολογίες. Οι προτάσεις που περιέχονται στο σχέδιο έκθεσης βασίζονται στην εξέταση που κάναμε του θέματος διαπιστώνουμε ότι μειώνονται οι αμυντικοί προϋπολογισμοί στα κράτη-μέλη και πρέπει να εξετάσουμε εάν για να προστατεύσουμε τους λαούς μας δεν θα έπρεπε να κάνουμε από κοινού ορισμένες προσπάθειες να επανεξετάσουμε τη λειτουργία των αγορών για θέματα άμυνας, να αποφύγουμε τον κατακαιρματισμό τους, να έχουμε δηλαδή μια βιομηχανική πολιτική στον τομέα της άμυνας με ευρωπαϊκή διάσταση. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή μας υπέβαλε μια θαυμάσια ανακοίνωση για το θέμα αυτό. Την ευχαριστώ. Χαιρετίζω την ανακοίνωση γιατί συμβάλλει στη συζήτηση για τις τροπολογίες τώρα που υπευλήθησαν από τους κοιόδης συζητητές αλλά και από πολλοί άριθμους άλλους ε, συναδέλφους τους οποίους ευχαριστώ. Υπάρχουν θαυμάσιες ιδέες σε αυτές τις τροπολογίες τις οποίες ε, φυσικά θα υποστηρίξω Διαβάζοντας όλες τις τροπολογίες ε, νομίζω ότι θα μπορούσα να καταλήξω σε συμβιβασμούς. Θα κάνω προτάσεις στους ε, σκιώδες συγητές. Ε, θα έχουμε μια συνάντηση την άλλη εβδομάδα στην παράγραφο 1. Εξετάζουμε ότι επειδή ο κόσμος αλλάζει, οι ευρωπαϊκοί λαοί που έχουν ένα κοινό πεπρωμένο πρέπει να προστατευτούν αλλά να έχουν τη δυνατότητα να παρεύουν στην διεθνή σκηνή και αξιοποιώντας την επιστημονική μας γνώση. Επειδή διαπιστώνουμε ότι πέρα από τις μεραρχίες και τους στρατιώτες είναι πολύ σημαντικές και οι επιστημονικές πλευρές ε, και η γνώση, μέχρι τα όρια της γνώσης. Υπάρχουν διαφορετικές ε, διατυπώσεις. Πιστεύω ότι μπορούμε να καταλήξουμε σε συμβιβασμούς γιατί σε όλες τις τροπολογίες δεν βλέπω να τίθεται ένα αμφιβόλο η γενική μου προσέγγιση. Στην παράγραφο 3 για τον κατακαιρματισμό της αγοράς. Ο Σνάλφος Βέμπερ πιστεύει ότι είναι καλύτερα να συνδυαστεί με την παράγραφο 4 και εδώ πιστεύω θα συμφωνήσουμε. Και τέλος, στην παράγραφο 11 που ε, ασχολείται με τη συνεργασία και τις κοινέ προσπάθειες και τονίζει τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Άμυνας. Ξέρουμε ότι δεν αξιοποιείται πλήρως και ότι είναι στη διάθεσή μας ο οργανισμός αυτός για να μας βοηθήσει με τη συμφωνία και των κυβερνήσεων και του Κοινοβουλίου μας ε, στην ε, διατύπωση και εφαρμογή πιο προωθημένων πολιτικών στον τομέα αυτό. Θα δούμε ποιες είναι οι κατευθύνσεις που θα μας δώσουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων. Όπως είπα και στους κοιόδης συγητές, στην έκθεσή μου δεν θα ασχοληθούμε με την ε, χρηματοδοτική πλευρά του θέματος. Ειλικρινά σας λέω, όλοι μαζί αποφασίσαμε να μην μιλήσουμε για δαπάνες είπα στο Μίχαελ Γκάλερα και συμφωνήσαμε ότι σε τέλος θητείας ε, τα οικονομικά θέματα είναι τόσο δυσμενή. Ε, μιλήσαμε για τον ορίζοντα 2020. Ο Κριστιαν Έλερ σωστά είπε ότι δεν συμπεριφέρεται σωστά εναντί μας στο Συμβούλιο. Ε, είναι πολύ σημαντικό θέμα, αλλά δεν θα το συζητήσουμε τώρα αυτή τη στιγμή. Δεν θελήσαμε λοιπόν να ασχοληθούμε με την χρηματοδοτική πλευρά. Η πρόταση που κάνουμε και που δεν είναι γραπτή βέβαια είναι να το συζητήσουν οι πολιτικές ομάδες στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας ακριβώς για τις εκλογές ε, του 2014 και επειδή θα αναθεωρηθεί ο προϋπολογισμός το 2016 να αξιοποιήσουμε τότε την ευκαιρία εάν στις εκλογές καταδειχθεί ότι οι λαοί συμφωνούν με τις κατευθύνσεις που τους, προτάν, που τους προτείνουμε με βάση τις κατευθύνσεις του Κοινοβουλίου μας, της Επιτροπής των Αρχικών Κρατών και Κυβερνήσεων, τότε λοιπόν θα επανεξετάσουμε τη δημοσιονομική πλευρά. Είναι κάτι θελημένο λοιπόν. Ο κύριος Γκέρεκ στην τροπολογία 51 προτείνει κάτι πρωτότυπο να δημιουργήσουμε ένα Ινστιτούτο Άμυνας και Ασφάλειας στα πλαίσια του κοινού κέντρου έρευνών. Πολύ καλή ιδέα. Ξέρετε, αν δούμε την ε, ευρωπαϊκή ιστορία, βλέπουμε πόσοι πόλεμοι έγιναν, πόσοι εμφύλοι, πόσοι θρησκευτικοί πόλεμοι. Διαπιστώνουμε λοιπόν ότι προχωράει η έρευνα και η επιστήμη γιατί χρειάζονται οι λαοί την έρευνα της επιστήμης. Πρέπει και σε περίοδο ειρήνης λοιπόν να συνεργαζόμεθα η δημιουργία ενός Ινστιτούτου στα πλαίσια του Κοινού Κέντρου Ερευνών που να εξετάζει τις πιο προωθημένες επιστημονικές ιδέες και να αναπτύσσει την επιστήμη μου φαίνεται ιδιαίτερα σκόπιμη. Τέλος, για την τελική παράγραφο που είναι οι συστάσεις προς το, Ευρωπαϊκό Συμβούλιο γιατί προς, αυτήν προς αυτό το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο απευθυνόμεθα όχι ως συνήθως προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα επιδιώξω μια συνενετική διατύπωση να ζητήσουμε δηλαδή από τους αρχηγούς κρατών και κυβερνήσεων να στηρίξουν πολιτικά στο υψηλότερο επίπεδο την προσπάθεια δημιουργίας επιστημονικής και τεχνολογικής βάσης για την Ευρωπαϊκή Άμυνα. Καταλήγοντας, ευχαριστώ ιδιαίτερος όλους ε, εκείνους με τους οποίους συνεργάστηκα, τους συνεργάτες μου, την κυρία Κολέ, τον κύριο Βαναρό και όλους τους άλλους ε, υπαλλήλου που με βοήθησαν και βεβαίως θα σας ακούσω για να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμβασμούς. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Οντή για την εισαγωγική παρουσίαση. Οι τώρα, ο κύριος Γκυρέκ, η κυρία Βαλιάν και ο κύριος Πρόντι. Αν θέλουν και άλλοι συνάδελφοι να εγγραφούν στον κατάλογο, παρακαλώ, ας το δηλώσουμε τώρα. Ευχαριστώ. Συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Οντή ως προς τις συστάσεις του. Υποστηρίζω και τις τροπολογίες που έχει καταθέσει. Βλέποντας ε, τις θέσεις των πολιτικών ομάδων δεν θεωρώ ότι θα υπάρξουν ε, αμφιλεγόμενα ζητήματα. Η Ευρώπη όντως έχει ε, γίνει μουσείο στον τομέα της άμυνας διότι ε, για υπερβολικά μεγάλο χρονικό διάστημα τελούσαμε υπό την αιγίδα των ΗΠΑ και ξέρουμε ότι εσχάτως ε, άλλαξε το προφίλ της και το αναπροσανατόλησε τις δράσεις της ε, η Αμερική προς τη Μέση Ανατολή και την Ασία. Δεν μπορούμε όμως να αφήσουμε αθωράκιστη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η προστασία της ειρήνης σημαίνει ότι προετοιμάζει κάποιος το αμυντικό του σύστημα με καινοτόμο τρόπο, με σύγχρονο τρόπο βάσει των νέων διαθέσιμων τεχνολογιών. Είναι σίγουρο λοιπόν πως ε, ο αμυντικός μας εξοπλισμός πρέπει να εξυγχρονιστεί. Ε, είναι προφανές ότι πάντοτε ελοχεύει κίνδυνος, ε, κυρίως μεσούσης της κρίσης, Πολλά κράτη-μέλη αποφασίζουν και εφαρμόζουν περικοπές των αμυντικών τους δαπανών. Η Πολωνία, παραδείγματο χάρη, η χώρα μου, που μέχρι τούδε ξόδευε 2% του ΑΕΠ για τις αμυντικές δαπάνες, που είναι υψηλό ποσοστό και πιστεύω ότι αυτό θα έπρεπε να είναι το ποσοστό και για άλλες χώρες. Ακόμη λοιπόν και η Πολωνία περιέκοψε τον αμυντικό της προϋπολογισμό λόγω των ευρύτερων δημοσιονομικών προβλημάτων που έχει. Δεν πιστεύω ότι είναι καλή λύση διότι και η πολωνική αμυντική βιομηχανία πρέπει να εξυγχρονιστεί, εξυγχρονιστεί και περιμένουμε ακόμη τις πρώτες ενδείξεις του εξυγχρονισμού αυτού. Οι προτάσεις που έχουμε καταθέσει, παραδείγματο χάρη, η πρόταση εναρμόνισης, για να το θέσω ευρέως, εναρμόνισης των ευρωπαϊκών αμυντικών βιομηχανιών, που δεν έχουν υιοθετηθεί προς το παρόν. Αυτές οι προτάσεις λοιπόν θα μπορούσαν να μας οδηγήσουν σε νέες συνεργατικές σχέσεις κυρίως για δράσεις χωρίς κόστος, θέσπιση προτύπων για, την, για ένα ομοιόμορφο αμυντικό σύστημα, ε, εισάγοντας πρότυπα για νέα είδη ε, αμυντικού εξοπλισμού Και παρόλα αυτά δεν είναι ρόδινα τα πράγματα, παρότι δεν συνεπάγεται αυτό επιπρόσθετο κόστος. Να σας δώσω ένα παράδειγμα. Όταν είχαμε τα προβλήματα στη Λιβύη, ξέρετε ότι προσγειώθηκαν εκεί πολύ καλά σουηδικά μαχητικά αεροσκάφη. Όταν όμως χρειάστηκε να επαναπατριστούν, απεδείχθη ότι δεν μπορούσαν να τροφοδοτηθούν σε καύσιμο διότι το είδος ε, καυσίμου στη Λιβύα διέφερε σε τέτοιο βαθμό από το είδος καυσίμου που χρησιμοποιούσαν που δεν ε, ήταν αδύνατη, αδύνατος ο ανεφοδιασμός τους. Το ίδιο και για τους οπλικούς μηχανισμούς. Το διαμέτρημα πρέπει να είναι ομοιόμορφο και διαλειτουργικό ε, για να μπορέσουμε να αλληλοβοηθούμαστε αν ε, συντρέξει ανάγκη. Ο κύριος Σοντή ε, ανέφερε επίσης ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό να δημιουργήσουμε ένα κέντρο, ένα Ινστιτούτο στα πλαίσια του Κοινού Κέντρου Ερευνών για ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση στον τομέα της άμυνας. Ένα τέτοιο Ινστιτούτο θα μπορούσε να βασιστεί στις νέες σύγχρονες τεχνολογίες και γιατί όχι, εν ευθέτω χρόνο, το Ινστιτούτο αυτό θα μπορούσε να επεξεργαστεί και την ε, αντιπυραυλική ασπίδα. Είναι πάρα πολύ καυτό το ζήτημα στην Πολωνία. Θα ήταν πάρα πολύ χρήσιμο να, να προ, μπορέσουμε να ε, της χώρες μας λαμβάνοντας υπόψη και το διαστημικό σκέλος, γιατί κάποιοι πύραυλοι πλέον μπορούν να εκτοξεύονται με αυτόν τον τρόπο, εάν βεβαίως κάποιος στον κόσμο στον οποίο ζούμε πάρει τέτοιες παράλογες αποφάσεις. Πρέπει όμως ε, να εξετάσουμε τέτοια σενάρια. Η Βόρειος Κορέα, παραδείγματος χάρη, διαθέτει τέτοιους πυράβλους και μπορούν να εκτοξευθούν κατά τη ΣΥΠΑ ή και το αντίστροφο είναι πάρα πολύ ε, το ζήτημα και οι υπουργοί μας θα έπρεπε να αφιερώσουν λίγο χρόνο για τη συζήτηση αυτή. Κλείνοντας. Να προσθέσω ότι θα έπρεπε να κρούσουμε τον κόδωνα κινδύνου στους υπουργούς που θα συσκεφθούν το Δεκέμβρη κατόπιν ετοιμάτως του Πρόεδρου Φανερόμπεϊ διότι θα, χρειαστεί να συζητήσουν αυτή την ε, αμυντική πολιτική. Και ένα λεπτάκι θα ήθελα να προσθέσω και κάτι για τον κύριο Ντί. Θα ήθελα να έχουμε το ταχύτερο δυνατόν του τροπολογίε σε όλες τις γλώσσες. Ε, ο κύριος Τσίτσεστερ, ναι, η γραμματεία θα τον φροντίσει. Ε, η κυρία Βαλέαν. Ευχαριστώ τον εισηγητή. Πολύ καλή έκθεση. Από πλευρά τη ομάδα των φιλελευθέρων. Έχω συνυπογράψει κάποιε από τι τροπολογίε. Η προσέγγιση νομίζω είναι ισορροπημένη. Προσπαθεί να λάβει υπόψη τις ανάγκες άμυνας, τις ανάγκες της βιομηχανίας, τις ιδιομορφίες. Οι τροπολογίες μας ε, τονίζουν τη σημασία της στρατηγικής αυτονομίας ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης, χωρίς βεβαίως να αποθαρρύνουμε τη συνεργασία γιατί βοηθάει την ανάπτυξη της τεχνογνωσίας, τις ανταλλαγές λοιπόν με τους εταίρους μας. Επίσης, θέλουμε να υπάρξει περισσότερη αμοιβαία διαφάνεια, γιατί έτσι θα αποφύγουμε τις επικαλύψεις, ε, το πρόσθετο κόστος και θα βοηθήσει γενικότερα την ενίσχυση της ασφάλειας. Θέλουμε να εναρμονιστούν οι κανόνες και οι προδιαγραφές γιατί έτσι θα είχαμε περισσότερο ανταγωνισμό στην ε, ενιαία αγορά παρά το ότι είναι πολύ ευαίσθητος και λεπτός αυτός ο τομέας. Συμφωνώ επίσης πολύ με τον εισηγητή που ε, είναι υπέρ της διτής χρήσης των τεχνολογιών και των προϊόντων, ειρηνικής και στρατιωτικής δηλαδή. Επίσης, οι αναδυόμενες οικονομίες ε, κάνουν όλο και μεγαλύτερες επενδύσεις ε, στον τομέα αυτό. Άρα η έρευνα και ανάπτυξη και η καινοτομία πρέπει να συνεχίσει να είναι μέλημά μας είναι πολύ καλή λοιπόν η έκθεση αυτή και θα συνεργαστούμε για να υποβάλουμε στο Συμβούλιο ένα πραγματικά ρωμαλαίο κείμενο. Ευχαριστώ πολύ ο κύριος Τσίτσεστερ. Και τώρα ο κύριος Πρόντι. Ευχαριστώ πολύ πρώτα απ' όλα τον συνάδελφο Οντί για αυτή την έκθεση Πρέπει να πω όμως ότι ε, δεν είμαι καθόλου ικανοποιημένος, όχι από την έκθεση βέβαια, αλλά από τη γενικότερη κατάσταση. Ας μην κρυβόμαστε πίσω από το δάχτυλό μας. Δεν είναι δυνατόν να μιλάμε για άμυνα και για αμυντικό υλικό χωρίς να έχουμε ταυτοχρόνως και μια κοινή πολιτική άμυνας. Ε, παράδειγμα τρανό είναι η Airbus. Υπάρχει λοιπόν μια επιχείρηση που είναι ανταγωνιστική σε παγκόσμιο επίπεδο και για την ώρα δεν ε, έχει βρεθεί κάτι τέτοιο. Γιατί δεν είναι σαφώς προδιαγραμμένος ο ρόλος των, ε, του στρατού. Και υπάρχουν ομάδες, εθνικές ομάδες συμφερόντων οι οποίες αντιτίθενται σε οποιαδήποτε εξέλιξη του ζητήματος. Οι Ηνωμένε Πολιτείε έχουν ένα εκατομμύριο 200.000 στρατευμένους. Εμείς έχουμε δύο εκατομμύρια. Και η διαφορά λοιπόν είναι μεγάλη. Αυτό είναι θέμα ουσίας και πρέπει να υπογραμμιστεί. Και πρέπει να το μελετήσουμε. Ή θα βρούμε μία κοινή πολιτική ή, εν πάση περιπτώσει, να σταματήσουμε να μιλάμε για κοινή βιομηχανία, κοινή αμυντική βιομηχανία. Θα ήθελα επίσης να υπογραμμίσω τα εξής. Υπάρχουν και ε, κατασκευές ε, οι οποίες ε, μπορεί να έχουν χρήση και πολιτική και στρατιωτική και οι οποίες θα πρέπει να αναπτυχθούν περαιτέρω. Και αυτό το ενδεχόμενο ανταγωνισμού για, τις, για την μη στρατιωτική χρήση και γι' αυτό μπορεί να έχουμε μια εξέλιξη τύπου Airbus. θα πρέπει να το διερευνήσουμε. Είναι μια οδός λοιπόν προς διερεύνηση και οπωσδήποτε οφείλουμε να τονίσουμε την ανάγκη να αναπτυχθεί μια τέτοια ε, δραστηριότητα. Αυτή τη στιγμή έχουμε μπροστά μας σε μια μεγάλη πρόκληση όσον αφορά την άμυνα. Ε, ε, πρόκληση η οποία σχετίζεται με τον κυβερνοπόλεμο. Και αυτό δεν θα πρέπει να το παραβλέψουμε. Γιατί η μεγαλύτερη πρόκληση που έχουμε μπροστά μας είναι τούτη εδώ. Νομίζω ότι οι πόλεμοι πλέον θα ξεκινούν από τον κυβερνοχώρο. γιατί μπορεί κανείς να πετύχει το στόχο του με πολύ λιγότερο κόπο και πολύ λιγότερα έξοδα από ό,τι χρησιμοποιώντας τα, τα συμβατικά αμυντικά συστήματα. Ευχαριστώ. Thank you very much, Mr. Ευχαριστώ κύριε Πρόντι. Καλό είναι που προεδρεύω γιατί αλλιώ ε, πολύ θα ήθελα να συζητήσω μαζί σας αλλά συμφωνώ για τους κυβερνοπολέμους Εφόσον δεν έχουν ε, άλλοι συνάδελφοι ζητήσει το λόγο, να καλέσω την κυρία Κάιν Τζούμπερ από την Επιτροπή. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Η κυρία Στάιν Γούμπερ ε, ε, δεν είναι εδώ. Ε, μήπως μπορείτε να της δώσετε πέντε λεπτά για να έρθει. Um, Ευχαριστώ την Επιτροπή που δεν μακρηγόρησε. Κύριε Οντή, παρακαλώ θέλετε να κλείσετε τη συζήτηση. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ε, θαυμάσια προεδρεύεται με αξιοσημείωτη ταχύτητα. Ευχαριστώ τους συναδέλφους που πήραν το λόγο. Αγαπητέ συνάδελφε Γκέρεκ, βέβαια δεν θα συμφωνούσα ότι είμαστε μουσεία, είμαστε μουσείο ως ε, Ένωση, γιατί υπάρχουν ε, κράτη-μέλη που έχουν ε, αξιοσέβαστη στρατιωτική ικανότητα και αποτελεσματικότητα. Αλλά αυτό που είναι ιδιαίτερα ανησυχητικό για τους λαούς μας είναι η εξέλιξη της κατάστασης. Δηλαδή, οι αμυντικοί προϋπολογισμοί των κρατών μελών είναι βεβαίως ακριβοί και δυστυχώς πολύ συχνά περικόπτονται. Και κάποια στιγμή δεν θα έχουμε στις χώρες μας στρατούς που να είναι σε θέση να υπερασπιστούν τα σύνορά μας και αυτό είναι υποχρέωση των συνθήκων. Πρέπει να μας ανησυχεί αυτή η τάση και γι' αυτό ο Πρόεδρος του Συμβουλίου ζήτησε οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων να ασχοληθούν με αυτό το θέμα. Έχετε δίκιο, Σνάλφε Γκέρεκ. Πρέπει και εμείς να εξετάσουμε κατά πόσο είμαστε ακόμη ανεξάρτητοι. Τώρα δεν θα μιλήσω για τα θέματα κατασκοπίας που ιδιαιτέρως μας στενοχώρησαν από πλευράς των ΗΠΑ αλλά επειδή είναι δημόσια η συνεδρίασή μας πρέπει να χαιρόμαστε που έχουμε το σύστημα Γαλιλαίος. Μας κόστισε 30 δορυφόρους. Το Κοινοβούλιο έσωσε το Γαλιλαίο και σήμερα διαπιστώνουμε ότι έχουμε δίκιο που έχουμε τις δικές μας τηλεπικοινωνίες. Το δικό μας σήμα ανεξαρτήτως των ΗΠΑ. Τότε είχαμε πει φανταστείτε τι θα γίνει αν υπάρξει ε, ένα στρατιωτικό ατύχημα και οι Ηνωμένε κόψουν τις τηλεπικοινωνίες, ε, τις δορυφορικές τις δικές τους. Τώρα έχουμε τις δικές μας. Έχουμε και σύστημα GPS δικό μας. Θυμάμαι τότε τι είχε πει ο Τζο Μπάιντεν. Είχε έρθει το 2010 εδώ στο σώμα μας και τι είπε η Αμερικανική κυβέρνηση θα είναι πολύ διαφορετική από τις προηγούμενες να έχετε υπόψη ότι η Αμερική δεν θα μπορεί να τα κάνει πια όλα Βεβαίως εσείς οι Ευρωπαίοι έχετε διεθνή ρόλο, αλλά θα πρέπει να ασχοληθείτε με τις γειτονικές σας περιοχές. Επιτέλους, για την προστασία, την ευημερία, την ειρήνη, την ασφάλεια, πρέπει να ασχοληθούμε με τα θέματα αυτό, αυτά και κυρίως με τη βιομηχανία και την επιστημονική έρευνα. Κυρία Βαλεάν, σας ευχαριστώ για την υποστήριξή σας, για τις τροπολογίες σας. Κάποια θέματα ανταγωνισμού πρέπει να τα συζητήσουμε γιατί κάποιες ε, τροπολογίες των σοσιαλιστών για τις ε, βιομηχανίες όπλων ε, πρέπει να δούμε πώς ακριβώς θα τις συζητήσουμε για να καταλήξουμε σε συμβασμούς αλλά γενικά σας ευχαριστώ για τη στήριξή σας. να είστε πρώτοι, έχετε δίκιο. Η τρέχουσα κατάσταση δεν μας ικανοποιεί αλλά πρέπει να πω υπέρ των κρατών μελών ότι τα στρατιωτικά θέματα είναι θέματα εθνικής κυριαρχίας. Είμαστε σε φάση οικοδόμης της Ευρώπης. Άρα, έχουμε την εξή σειρά. Προπαρασκευαστική πολιτική συζήτηση. Την έκανε η Κομισιόν για να εκπονήσει την ανακοίνωση. Θα την κάνει το Συμβούλιο. Θα την κάνουν οι πολίτες στα πλαίσια της προεκλογικής εκστρατείας για τις εκλογές του χρόνου. Αυτή λοιπόν η διαδικασία πολιτικής αναζήτησης πρέπει να οθήσει την Υπηρώ μας, να οργανώσει καλύτερα, να διανύμει καλύτερα, να μοιραστεί καλύτερα για να αποφασίσουμε από κοινού για τις ε, βιομηχανικές ε, και ερευνητικέ πλευρές της άμυνας θέλουμε να συνεργαστούμε. Η χώρα μου έχει μία συμφωνία συνεργασίας με το Ηνωμένο Βασίλειο για την ε, στρατιωτική συνεργασία και την έρευνα στον τομέα αυτό που την είχε συνάψει η προηγούμενη κυβέρνηση. Απευθύνθηκα στη σημερινή κυβέρνηση. Του είπα τι θα κάνετε και απάντησαν βεβαίω. Θα συνεχίσουμε να την εφαρμόζουμε. Πολύ καλή ιδέα να συνεχίσουμε τη συνεργασία. Δεν έχουμε πια τη δυνατότητα ο καθένα να τα κάνει μόνο του. Έχουμε λοιπόν ήδη πείρα από τέτοιε συνεργασίε Πρέπει λοιπόν να συνεργαστούμε, να το συζητήσουμε. Δεν είμαστε κατά των Αμερικανών, δεν σημαίνει κάτι τέτοιο. Ήρθε η ώρα να αναλάβουμε την ευθύνη της προστασίας μας, να δούμε τι μπορούμε να κάνουμε μαζί, για να μοιραστούμε και τις δαπάνες, για να αυξήσουμε την αποτελεσματικότητα και για να εφαρμόσουμε τις αξίες μας. Η πρώτη μας αξία είναι η ειρήνη, πήραμε το βραβείο Νόμπελ ειρήνης, για να υπάρξει όμως ειρήνη όπως μας αποδεικνύει η παγκόσμια κατάσταση, πρέπει να είμαστε έτοιμοι για πόλεμο. Οι στρατιωτικές πλευρές είναι λοιπόν ένα θέμα που πρέπει να μας απασχολήσουν. Όλες οι πολιτικές ομάδες πρέπει να συμβάλλουν με τις απαντήσεις τους και χαίρομαι που οι ομιλίες και οι τροπολογίες σας μοιάζουν να δείχνουν ότι υπάρχει συνένεση για την βιομηχανική βάση και την επιστημονική έρευνα ε, μίλησα πολύ για να δούμε μήπως ε, θα φτάσει η Κομισιόν αλλά η Κομισιόν δεν ήρθε, δεν έχω τίποτα άλλο να πω δεν ξέρω τώρα τι θέλετε να κάνουμε να συνεχίσω Πρόεδρος Μα πότε δεν θα ήθελα να αποθαρρύνω τους συναδέλφους ε, από το να πάρουν το λόγο. Αλλά αν είπατε ότι είχατε να πείτε, μπορείτε να σταματήσετε να μιλάτε. Ήταν πολύ ενδιαφέρουσα η συζήτηση. Σας ευχαριστώ για την ε, ομιλία σας. Οπότε, να υπενθυμίσω σε όλους ότι η ψηφοφορία για την έκθεσή σας στην Επιτροπή μας θα γίνει 7 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο. Θα συνεδριάσουμε για ε, ε, αρκετές ώρες τη Δευτέρα το βράδυ. Πολύ μας χαροποιεί αυτό σίγουρα. Είναι η επόμενή μας συνάντηση. Διάφορα. Έχουμε μια κοινή συνάντηση της Επιτροπής μας και των συνεργατών μας στην Επιτροπή Περιβάλλοντος ε, το σήμερα το απόγευμα στις 3. Ε, στο πλαίσιο για το περιβάλλον 2030 θα εκπροσωπηθεί και η Επιτροπή μας. Αυτά, υπό τα διάφορα δεν βλέπω να υπάρχει τίποτα. Λύεται τη συνεδρίαση. Θα τα πούμε στην επόμενη συνεδρία. Σας ευχαριστώ.